Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Το πρώτο θέμα αφορά την Κένια και την αποτυχία σύλληψης του Προέδρου Ομάρ Αλ Μπασίρ. Και ο πρώτος που θα λάβει το λόγο επ' αυτού είναι ο κύριος Τάνο για 1,5 λεπτό. Ο πρόεδρος Μπασίρη κατηγορείται για γενοκτονία από το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, διότι φέρονται και ε, διαπράξει εγκλήματα στον Ταρφούρ. Οπότε, πώ να θεωρήσουμε ότι είναι τιμόμενο προσκεκλημένο. Ε, τον ε, κάλεσε πέρσι η Τουρκία, δεν τον κάλεσε η Τουρκία στο, στη σύνοδο της Άγγελας πέρσι και όπως είπε ο, ο πρόεδρος της Κένιας, ευκαιρία το νέο σύνταγμα της χώρας ε, είπε ότι υπάρχουν διάφοροι υπουργοί εκεί και ο Πρωθυπουργό Ντίγκα και άλλοι στην ευάλωτη κυβέρνηση ανησυχούν για, την παρουσία του Μπάσιρ. Όμω το, η ζημιά έγινε και ε, το, το, το, αμαυρώθηκε η χώρα γιατί ακριβώς ε, έκρινε ότι είναι δυνατόν ακόμα και αρχηγοί κρατών να δικαστούν από το δικαστήριο αυτό, ιδίω για τέτοια εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα, εγκλήματα πολέμου, γενοκτονίε και το επομένω ότι έχει την δοσηδικία, την αρμοδιότητα και την περίπτωση, αλλά η Κένια δεν δέχθηκε να το κάνει αυτό, παρά το έχει προσυπογράψει να είναι μέλο του ICC, του δικαστηρίου αυτού. Οπότε θα πρέπει να διερευνήσουμε επίση και όλα αυτά τα οποία έγιναν στι εκλογέ, η Δοβία δηλαδή πριν από τρία χρόνια και ε, επομένως αυτό έρχεται σαν εξέλιξη των προβλημάτων που είχε χώρα τότε με τις εκλογές. Σάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Η Κένια είναι τέρος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη, εμπόριο κλπ. Και ήταν ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου προσυπέγραψε την τέταρτη πράξη όσον αφορά την Αφρικανική Ένωση και έχουμε συνάψει συμφωνία όπου ορίζονται οι όροι της εταιρική μας σχέσης. Και επομένως οι ενισχύσει μας προς αυτή τη χώρα προϋποθέτουν τήρηση των υποχρέωσεων της χώρας. Έγινε όμως στις 27 Αυγούστου ο Μάρας Μπασίρ επισκέφθηκε σαν επίσημος προσκεκλημένος της κυβέρνησης στη χώρα. Και αυτό έγινε παρά το ότι υπήρχε ένταλμα Δίωξη εναντίον του λόγου των εγκλημάτων που το διαπραξίες στο Νταρφούρ. Θα πρέπει επομένω να προσαχθούμε του Διεθνού Δικαστηρίου, αλλά η Κένια υποχρεούται να τον συλλάβει. Δεν το έπραξε. Είναι σοβαρό το πρόβλημα και είναι ένδειξη ότι η κυβέρνηση της χώρας δεν είναι αξιόπιτη όσον αφορά τις διεθνείς της ανηλυμένες υποχρεώσεις και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα να εξασφαλίσουμε επομένω ότι δεν θα υπάρξει ατιμορρησία. Και επομένω αν κάνουμε κάτι και εμείς οι ίδιοι θα είμαστε συνεπείς όσον αφορά τη βοήθειά μας προς την Αφρική να έχει δημοκρατία και σταθερότητα. Παρακαλώ ο υψηλό εκπρόσωπο να αναλάβει διπλωματικέ συνέργειας έναντι της ε, για να τι ε, υπενθυμίσει τι υποχρεώσει τη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. δυόμιση λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, στο συνέδριο φέτος στην Καμπάλα για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατέστη σαφές πώς θα λειτουργήσει αυτό το δικαστήριο μόνο αν το υποστηρίξουν τα κράτη, ειδικά αυτά τα οποία επικύρωσαν το καταστατικό της Ρώμης και τα κράτη-μέλη της Ένωσης πρέπει να το θυμούνται, γιατί συχνά ο φόβος διπλωματικών περιπλοκών και πολιτικών περιπλοκών εμποδίζει την συνεπή δράση όπως παραδείγματο χάρη την σύλληψη υπόπτων για εγκλήματα πολέμου. Στη σημερινή συνεδρίαση ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση της Κένιας που προσκάλεσε τον Ομάρα Αλμπασίρ και δεν τον συνέλαβε. Υπάρχουν εντάλματα εις βάρος του Αλμπασίρ για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου. Άρα η Κένια παρεμβίασε το διεθνές δίκαιο και τίμησε την λεγόμενη αφρικανική αλληλεγγύη η οποία είναι ισχυρότερη από το διεθνές δίκαιο σε περιπτώσεις ακόμα και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για τα εκατομμύρια Αφρικανών που υπέφεραν από τις φρικαλαιότητες του Προέδρου Μπασίρ και από άλλους εμφυλίους πολέμους στην Αφρική. Τα θύματα και οι συγγενείς τους χρειάζονται δικαιοσύνη, πρέπει να δουν αυτόν τον αυτούς τους εγκληματίες να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους όσο υψηλά ιστάμενοι και αν είναι. Πρέπει επίσης να ασκήσουμε κριτική στο ότι και η Αφρικανική Ένωση είναι κατά της σύλληψης του Ομάρ Αλμπασίρ και λέει είναι υπέρ αυτής της λανθασμένης αλληλεγγύης και έτσι εξασθενεί την τόσο απαραίτητη ορθή διακυβέρνηση, μια ορθή διακυβέρνηση η οποία θα τηρεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Επίση. απογοητευτικό είναι πω αρνήθηκε η Αφρικανική Ένωση να συστήσει περιφερειακό ποινικό δικαστήριο στην Αντίσα Μπέμπα. Πρέπει η Κομισιόν να δει αυτή τη μη συνεργασία έναντι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να το βάλει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Συνόδου Κορυφής με την Αφρικανική Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Βέζια για 2,5 λεπτά. Στο είμαστε αρκετοί που λυπούμεθα για την απόφαση της Κένια και της, ε, του Αραβικού Συνδέσμου να μην εφαρμόσουν ε, το, την, ε, την, το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Ομάρ Αλμπασίρ στην ουσία χέρι ασυλίας ο Μπασίρ στο σύνολο των Αφρικανικών και Αραβικών χωρών. Εμείς θα θέλαμε η διεθνής δικαιοσύνη να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους και για όλους σε όλο τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο δρόμος είναι μακρύς έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ουσιαστικά το δικαστήριο αυτό. Θα ήμασταν πιο αξιεπιστοί αν περισσότερες χώρες όπως η Γαλλία δεν καθυστερούσαν στην προσαρμογή της οικονομίας τους και γενικότερα γενικότερα των νομικών του συστημάτων ε, στο σύστημα το οποίο επιβάλλει πλέον το διεθνές ποινικό. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μεγάλες ευθύνες απέναντι στην Αφρική και δεν θα πρέπει να τους δώσουμε την εντύπωση δύο μέτρων και σταθμών. Η διεθνής δικαιοσύνη φαίνεται ότι εφαρμόζεται κυρίως στις αφρικανικές χώρες, εκτός αν οι κυβερνήσει ορισμένων χωρών της Ευρώπης έχουν τοπικά υψηλά συμφέροντα. Λυπούμεθα λοιπόν που η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου δεν εφαρμόστηκε για τον Μπασίρ που είναι υπεύθυνο για σειρά εγκλημάτων. Θα θέλαμε όμως να εφαρμόζεται στο σύνολο των χωρών του κόσμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ένας πραγματικός χώρος ελευθερίας και δικαιοσύνης και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην καθολική εφαρμογή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σήμερα το πρωί μια μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδίκασε τις διακρίσεις εις βάρος του Ρομ και τις ξενοφοβικές ιδέες του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας που αναφέρθηκε ότι θράσος στην διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν τα λόγια μας να γίνουν πράξη. Μπέρμαν δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν λίγοι λόγοι να πιστεύουμε στην πρόοδο. Φαίνεται πως και σε αυτό τον αιώνα θα εξακολουθήσουμε να έχουμε πολέμους και απρότητες. Εάν υπάρχει ένα βήμα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ξεκίνησε με το Δικαστήριο της Ιουγκοσλαβίας, μετά της Ρουάντας και οδηγηθήκαμε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν θα ήταν ένα δικαστήριο των νικητών όπως αυτό της Νιρεμβέργης, αλλά ένα ανεξάρτητο δικαστήριο που θα απέδιδε δικαιοσύνη και βεβαίως τα κράτη θα πρέπει από μόνα τους να εφαρμόσουν τις συνθήκες που έχουν υπογράψει. Έτσι μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη διεθνή ειρήνη, να μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση και να ικανοποιηθούν τα θύματα. Χάρη σε αυτό το δικαστήριο οι μελλοντικοί ε, εγκληματίες πολέμου θα μπορέσουν να λογοδοτήσουν καθώς δεν επιτρέπεται και δεν είναι δυνατό να υπάρχει ατιμορρησία και οπωσδήποτε όχι στην περίπτωση ο Μάρα Αλμπασούρ. Η Κένια υπέγραψε το καταστατικό της Ρώμης και βεβαίως πάκτα στον Σερβάντα οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται. Οπότε το να λειτουργεί να κυκλοφορεί ανεμπόδιστο στην Κένια και να εορτάζεται η δημοκρατία μάλιστα ο Μάραλ Αλμπασίρ είναι κάτι το ανησυχητικό. Θα ήθελα και εγώ όπως και η συνάδελφος να απευθύνω έκκληση στις χώρες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει ακόμα το καταστατικό της Ρώμης. Τι περιμένει πια ο Μπαράκ Ομπάμα. Θεωρούμε λοιπόν πως θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια παγκοσμία τάξη η οποία δεν θα αφήνει ατιμόρυτους εγκληματίες πολέμου οπουδήποτε και αν είναι στον κόσμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Κέλαμ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα που σήμερα συζητούμε είναι να δούμε τι γίνεται εφόσον η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη όσον αφορά τα νύχτα της ανθρωπότητας διότι κατηγορείται ο πρόεδρος Μπασίρ για τέτοιου είδους εγκλήματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και κρεμούν εντάλματα συλλήψεως εις βάρος του. Σήμερα το θέμα είναι το κατά πόσον υπάρχει η απαραίτητη βούληση αλλά και ο συντονισμό, ούτω ώστε οι κατηγορούμενοι αυτοί να προσάγονται από τις δικαιοσύνη. Στι 27 Αυγούστου η κυβέρνηση τη Κένια έχασε την ευκαιρία να το κάνει αυτό. Ε, ε, ε διότι τον εκάλεσαν τον Μπασίρο σε επίσημο προσκεκλημένο και ευτυχώ γνωρίζουμε ότι ο πρωθυπουργό τη χώρα παρεδέχθη ότι πρόκειτο περί λάθος και παραβίασης των δεσμεύσεων των διεθνών της χώρας. Ε, σήμερα θέλουμε έκκληση στις χώρες της Αφρικανικής ε, Ένωσης τόσο ώστε να ενώσουν τις πρόθειές τους με τη διεθνή κοινότητα και να προσεχθεί ενώπιον του δικαστηρίου ή στην Χάγη ο πρόεδρος Μπάσερ. Και εκεί βεβαίω θα έχει τα δύο κάθε κατηγορουμένο εις, ε, την εισπεράσπιση και χαιρόμαστε πάρα πολύ το ότι όλοι εδώ πέρα συμφωνούμε και θέλουμε τελικά να προσαχθεί ενώπιον του δικαστήριου της Χάγης ο πρώτος Μπασίρ. Και τώρα οι αγορητές των πολιτικών ομάδων. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Κάτσμαρεκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εμείς έχουμε μία παροιμία στα πολομικά. Ο λίγον έγκυος δεν γίνεται και έτσι προσπαθεί να συμπεριφερθεί και η Κένια. Δηλαδή και προσκαλούμε τον Αλμπασούρ, από την άλλη έχουμε υπογράψει και το καταστατικό της Ρώμης. Ε, δεν γίνεται. Είτε καταδιώκουν τους εγκληματίες, είτε δεν τους καταδιώκουν και τους αφήνουν ήσυχους. Η προσπάθεια να αποδειχθεί πως μπορούν αυτά τα δύο να συμβιβαστούν δεν στέκει και τα επιχειρήματα των κενιατικών αρχών πως είναι γειτονικό κράτος και έπρεπε να τον καλέσουν, ε, δεν είναι σοβαρό και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της Κένιας. Οι αρχές των ε, κρατών που έχουν υπογράψει πρέπει να τηρούν ε, ορισμένες, ε, ορισμένους κανόνες. Δεν αντιλαμβάνομαι πως θα έπρεπε κανείς να διώξει αυτούς τους κλιματίες, αλλά δεν το κάνει. Ευχαριστώ. κυρία Γκέριγκερτε Οντενμπέργκ για ένα μισή λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ιστορία δείχνει πως ε, κάποτε και οι εγκληματίες πολέμου αντιμετωπίζουν την ε, δικαιοσύνη. Όταν ειδικά νομίζουν ότι έχουν ξεφύγει ο Άντολφ Φάιχμαν, μετά από 15 χρόνια έρευνα συνελήφθη στο Buenos Aires. Το ίδιο και με Σέρβους που έφυγαν στα χρόνια της δικαιοσύνης 13 χρόνια μετά από τον πόλεμο. Ανάλογη μοίρα περιετνημένη και τον Ομάρα Αλμπασίρ για τα όσα έχει κάνει στο Νταρφούρ γιατί είναι καταζητούμενος. Τι μπορεί να κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει. Πρώτα απ' όλα να ασκήσει πίεση σε όσους έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Ρώμης για να την εφαρμόσουν κατόπιν. Έχουμε τους εορτασμούς ε, στην ε, Κένια πηγαίνει ο άνθρωπος, παρίσταται με την ισχύα του και μετά φεύγει ίσχος. Δεν μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να δούμε και να εκμεταλλευτούμε την συμμετοχή της ΥΠΑ της εκπροσώπου και να οδηγηθούμε τελικά μέσω της Συμφωνίας του Κοτονού στην σύλληψη του Αλμπασέ. Σας ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους. Κυρία Ρίς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υποδοχή με ανοιχτές αγκάλες στον κύριο Μπασίρ καταδικάζεται από το ψήφισμά μας σήμερα. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε κάποιες βασικές αρχές. Η Κένια, όπως και άλλες χώρες, πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και θα έπρεπε να διευκολύνουν τη σύλληψη του Μπασίρ για εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία στον Ταρφούρ. Θυμίζω στον Ταρφούρ μιλάμε για 300.000 αθώους νεκρούς. Υπάρχουν και άλλες χώρες βέβαια οι οποίες έχουν λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο, στη Λιβύη, το Κατάρι, Σαουδική Αραβία. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να έχει μία πολιτική, την πολιτική της αυστηρότητας, γιατί η Αφροκανική Ένωση έδωσε οδηγίες στα κράτη-μέλη της να μην συλλάβουν τον πρόεδρο Μπασίρ. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Άστον να τονίσει ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα πρέπει να είναι βασικός άξονας της συζήτησης της επόμενης συνάντησης Αφροκανικής Ένωσης ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάσκα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ. Ακριβώς το ότι μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερο σε Ασία και Αφρική ο πρόεδρος μας δείχνει το, το ότι δεν έγινε τίποτα όσον αφορά το ένταλμα σύλληψης για τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητας. Βιασμοί, βασανιστήρια, γενοκτονίε, γενοκτονίες, ε, προετοιμασία εγκλήματος, ε, διάφορα εγκλήματα κατά τη περιουσίας και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι ηγέτες ε, κρατών που δεν σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανοχή αντί τέτοιων εγκλημάτων κατά του αμάχου πληθυσμού. Και ο Ρωβικός Σύνδεσμος και Ένωση των κρατών της Αφρικής ενώ έχουν προσυπογράψει σχετική υποχρεώση δεν την τηρούν και έτσι δεν προσάγει το νόμο της δικαιοσύνης ο πρόεδρος Μπασίρ. δεν είναι δυνατόν να γίνεται αντιμετώπιση κάποιας επανάστασης με τέτοια εγκλήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θεωρώ σωστό το να ενισχύουμε τις κυβερνήσεις αυτές που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να εξηγηθεί ότι το να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους είναι ασυμβίβαστο με το να ζητούν βοήθεια και εμείς να τους την παρέχουμε. Πρόκειται περί βαρβαρικών καθεστώτων που έτσι υπερασπίζονται. Άρα όχι άλλα χρήματα προς εκείνους που δεν συνεργάζονται με το Διεθνές Δικαστήριο. Κυρία Κόρχολα. Ως ε, μέλος ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα πρέπει ε, η Κένια να τηρεί τις δεσμεύσεις και αυτό σημαίνει βεβαίως την εκτέλεση των ενταλμάτων εις βάρος του Αλμπασίρ. Θα πρέπει λοιπόν να πραγματοποιήσουμε τα όσα αναφέρονται στο πνεύμα του διεθνούς δικαίου. Το 2007 υπεγράφει και μια συμφωνία ειρήνης ε, που θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί στην χώρα. Μια επανάληψη της καταστροφής όπως τον Ταφούρ δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα ποτέ ξανά. Βεβαίως ε, πρέπει να ασκήσουμε κριτική στην Κένια για την στάση της, ε, όμως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να εφαρμοστεί η ειρηνευτική συμφωνία και ειδικά οι εκλογές οι οποίες προβλέπονται για φέτος να γίνουν και να αρθεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ε, στο σόταν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πρέντα. Ο Μάραλ Μπασίρη προκάλεσε ακόμη μία φορά τη εθνική κοινότητα. Η κενιατική κυβέρνηση τον είχε καλέσει στον εορτασμό του συντάγματο και δεν τον συνέλαβε και μάλιστα στο όνομα της καλής γειτονία. Ε, αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Η Κένια είναι κράτος μέλος του καταστατικού της Ρώμης, οπότε έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ειδικά μετά την ε, απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 7. Είναι υποχρεωτικό πλέον να συνεργαστούν όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Ο Κενιάτς Πρωθυπουργός είπε πως δεν ήθελε να συνεργαστεί λόγω του ψηφίσματος Αφρικανικής Ένωσης. Και αυτό είναι ασύμβατο με το διεθνές δίκαιο. Θεωρώ πως τα κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης θα πρέπει να είναι τα πρώτα τα οποία θα παλεύουν για τέτοιες υποθέσεις όταν υπάρχουν αυτά τα φρικτά εγκλήματα σε αυτή την Ήπειρο. Ευχαριστώ κύριο Σόνικ τώρα. Ευχαριστώ. Πρέπει να εκφράσουμε σαφώς ε, την άποψή μας ε, και τη στάση μας εναντί της κενιατικής κυβέρνησης και να μην στηρίζουμε πλέον τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος Αλμπασίρ ε, καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να κυκλοφορεί ελεύθερος ενώ κατηγορείται για βασανιστήρια, βιασμούς, εγκλήματα πολέμου και να τον υποδέχονται κιόλας με τιμές. Η Κένια έχει υπογράψει το καταστατικό, είναι λοιπόν υποχρέωση αυτής της χώρας να συλλάβει αυτό το άτομο ή να εμποδίσει την είσοδό του στη χώρα. Εγώ είμαι υπέρ της στήρησης των υποχρεώσεών μας. Απευθύνω έκκληση σε όλα τα αφρικανικά κράτη που μπορούν να συλλάβουν αυτό το άτομα. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι εγκληματίες να μην βρεθούν στη Χάγη. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην διαδικασία του KTI. Έχουμε περισσότερα αιτήματα από τη χρόνο. Θα ακούσουμε λοιπόν έναν από κάθε πολιτική ομάδα και να πω πως από εδώ και μπρος θα ήθελα να τηρείτε τον χρόνο αλλιώς θα χτυπάω το σφυράκι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο κύριος Νίκολασιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλούμε για αυτή την εκδήλωση η οποία αφορούσε το σύνταγμα της χώρας. Ήταν το πιο σημαντικό γεγονός από τότε που η χώρα έγινε ανεξάρτητη δεκαετία του 60. Όμως αμαυρώθηκε για πάντα η επίσημη αυτή ε, εκδήλωση από την παρουσία του Μπασίρ ο οποίος κατηγορείται για εγκληματικές ανθρωπότητες, εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και η Κένια τον κάλεσε επομένως απέδειξε ότι δεν συμμορφώνεται με το όσο έχει συμφωνήσει και με το κράτος δικαίου και η στάση αυτή της ε, Κένιας σε σχέση με τις διανύσεις της υποχρεώσεις είναι κάτι το οποίο προβληματίζει γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει η Κένια να επαναλάβει το ότι θέλει να συμμορφώνεται με τις διεθνείς συμφωνίες ε, και με, τις, με τα κείμενα που έχει προσυπογράψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γκόμεσα. Το κοινοβούλιο αυτό, η Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών πρέπει να καταδικάσουν την πρόσκληση που απευθύναν οι αρχές της Κένια στον πρόεδρο Αλμπασίρ. Δεν σεβάστηκαν το διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Αλμπασίρ για εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας και για συμμετοχή σε γενοκτονία. Η Κένια, θυμίζω, έχει υπογράψει τη Συμφωνία της Ρώμης, έχει υπογράψει επίσης και τη Συμφωνία της Κοτονού και πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες. Οι αρχές της Κένιας στη συγκεκριμένη περίπτωση υπονόμευσαν τα συμφέροντα της ίδιας τους της χώρας γιατί δεν συμμετέχουν στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να καταπολεμήσει ε, καταστάσεις και περιπτώσεις εγκληματιών όπως το συγκεκριμένο πρόσωπο, τον πρόεδρο του Σουδάν. Ε, Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η γενοκτονία είναι ένα σοβαρό έγκλημα. Όσοι την διέπραξαν και όσοι την σχεδίασαν θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουν την ε, δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει στην ερχόμενη σύνοδο με την Αφρικανική Ένωση να θέσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα να το έχει πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που διώκονται και γίνονται γενοκτονίες και θα πρέπει να ερευνηθούν ε, αυτοί οι φόνοι. Το ότι υπάρχουν εντάλματα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σημαίνει πως πρέπει και να εκτελούνται και τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να ε, γίνει αυτό πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Τέλος και ο Σόμπερμαϊρ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Ενημέρωσης του ΟΗΕ υποστηρίζει από το 2004 την αρχιτεκτονική της Αφρικανικής Ένωσης και έχει δώσει 300 εκατομμύρια ευρώ 2004-2007. Μα όλα αυτά έχουν νόημα εάν ε, συνεισφέρει ενεργά εκεί όπου υπάρχουν κρίσεις στην Αφρικανική Ήπειρο, η Αφρικανική Ένωση αλλά βλέπουμε πως δεν υπάρχει μεγάλη συνεργασία και με τη Λιβύη υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια και εδώ πέρα δεν εκδίδεται και ο πρόεδρος ε, του Σουδάν. Κοιτάξτε, απλά πράγματα. Πρέπει χωρίς παρεξηγήσεις και καθόλου κομψά να τα πει η πατή εκπρόσωπος. Λεφτά θα δίνουμε εάν η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Thank you. the Commissioner Thank you very much, Madam President. Ευχαριστώ τώρα η Επίτροπος για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σύστημα της Ρώμης είναι βασικό μέσο της διεθνούς κοινότητας για να καταπολεμήσει την ατιμορρησία για τα σοβαρότερα εγκλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Νομίζουμε ότι η προώθηση του καθολικού χαρακτήρα των μέτρων και των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι κάτι το θετικό για το σύνολο της οικουμένης. Το σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα βοηθήσει την προώθηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στον κόσμο και θα πρέπει όλες οι χώρες να επικυρώσουν τη συνθήκη της ε, Ρώμης. Στη συνάντηση κορυφής τον Ιούλιο η Αφρικανική Ένωση ζήτησε από τα μέλη της να μην εφαρμόσουν, το, να μην ασκήσουν το ένταλμα αυτό, το ένταλμα σύλληψης. Και προσελκύθηκε ο Αλμπασίρ να είναι παρόν στις εορτές για το νέο σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κένια και οι δύο αυτές ενέργειες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά φαινόμενα. Θα πρέπει η Κένια να σεβαστεί τις ανηλυμένες της υποχρεώσεις σε διεθνές επίπεδο και να σεβαστεί επίσης και τις υποχρεώσεις της σε επίπεδο διεθνούς δικαίου όπως και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την Κένια να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στα πλαίσια του διαλόγου που προβλέπεται από το άρθρο 8. Έχει αποδείξει βέβαια η Κένια ότι είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό για θέματα εσωτερικά της Κένια και αυτό απεδείχθηκε από την επίσκεψη του γραμματέα του δικαστηρίου στην Κένια την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα τώρα με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπρόσωπος της Αντιπροέδρου Άστον εξέδωσε μία δήλωση εκφράζοντας την ανησυχία της για την ανικανότητα ή αδυναμία καλύτερα της Κένια να συλλάβει τον Αλμπασίρ. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε ε, μέτρα έτσι ώστε να μεταφερθεί η άποψή μας αυτή και πίσημα προς την κυβέρνηση και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής εκφράστηκε η άποψη το θέμα να τεθεί προς συζήτηση και στην επόμενη συνάντηση κορυφής Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε Χέντεγκαρντ. Έκλεισε πλέον η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει άμα το τέλος των συζητήσεων. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη